the wrong thing. Okay, so dear colleagues... Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με το εργαστήριο. Καλώς ήρθατε μετά το διάλειμμα για το γεύμα. Αγαπητά μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω σε αυτό το εργαστήριο. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαστήριο. Επικεντρωνόμαστε στην πρόληψη εμπορίας ανθρώπων Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε τόσο συχνά κατά νου και είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα. Έχει ως ε, στόχο να συναντηθούν όσοι λαμβάνουν αποφάσεις εκπρόσωποι Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με τον αντίκτυπο της μεταναστευτικής κρίσης ε, στην εμπορία ανθρώπων και να αξιολογήσουμε τις ανάγκες στις διάφορες χώρες και να δούμε ποια συστήματα πρόληψης και αρρωγής στα θύματα υπάρχουν. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Κομισιόν για την πρόοδο που έγινε, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, έκθεση του 2016, διαφαίνεται ότι τα εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων έχουν εκμεταλλευτεί την κρίση για να στοχεύσουν τους πιο ευάλωτους, κυρίως τις γυναίκες και τα παιδιά. Αν δούμε την έκθεση αυτή, μπορούμε να δούμε ότι μιλά αυτή η έκθεση για 15.800 θύματα από το 2013 ως το 2014 και μιλάμε για σεξουαλική εκμετάλλευση, εργατική εκμετάλλευση, εμπορία οργάνων. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και για τους πρόσφυγες και θα ήθελα να καλωσορίσω τη συνάδελφο από το γραφείο της συντονίστρης ΤΣΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, την κυρία Σακυλιάδου. Καλώς ήλθατε. Πριν να της δώσω το λόγο, πρέπει να πω και κάτι για τους κανόνες. Ξέρετε τους κανόνες. Σας ενημέρωσε ο κύριος Μωράες την πρώτη συνεδρίαση. Θα δοθεί ο λόγος σε δύο μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εναλλακτικά. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν δύο λεπτά στη διάθεσή τους. Και τώρα θα σας δώσω το λόγο. Έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, μπορείτε να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση αυτή. Λέγομαι Ζουσέ Κελιόδο και εκπρόσωπο το Γραφείο Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Η κυρία Βασιλιάδου είναι αρμόδια. Αυτή η θητεία θεσπίστηκε το 2000, αυτή η εντολή θεσπίστηκε το 2011 με την ε, υποχρέωση να παράσχει προσανατολισμό και στρατηγική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Η εμπορία ανθρώπων είναι σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ταυτόχρονα. Πρόκειται για μια διεθνή απειλή, μια διεθνική μορφή οργανωμένου εγκλήματος, η οποία ε, ουσιαστικά ενισχύεται από τη ζήτηση και από τα υψηλά κέρδη. Όπως είπε και η κυρία Έρνστ, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση πρόοδου που δημοσίευσε η Κομισιόν, για την περίοδο 2013 μέχρι το 2014 είχαμε περίπου 16.000 θύματα εμπορίας ανθρώπων καταγεγραμμένα. Αυτό σημαίνει ότι αυτά είναι τα θύματα που κατά κάποιο τρόπο ήρθαν σε επαφή με τις αρχές. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά υψηλότερος και γνωρίζουμε ότι τα στατιστικά μας στοιχεία δεν μπορούν πάντοτε να αντικατοπτρίσουν ουσιαστικά την νομοθεσία των ανθρώπων που είναι θύματα εμπορία, κυρίω στο σημερινό μεταναστευτικό πλαίσιο. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, το 65% των και θυμάτων είναι υπήκοοι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η εμπορία ανθρώπων υπήρχε πριν τη μεταναστευτική κρίση και θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά τη μεταναστευτική κρίση. Το γεγονό είναι ότι η σημερινή κατάσταση, η προσφυγική κρίση, ουσιαστικά κάνει πιο έντονη τον ευάλωτο χαρακτήρα των ανθρώπων αυτών η πιο διαδεδομένη μορφή εκμετάλλευσης ε, είναι η εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση και τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και κορίτσια. Ακολουθούν το 21% των θυμάτων για εκμετάλλευση στον τομέα της εργασίας. Τα περισσότερα θύματα εκεί είναι άνδρες και αγόρια. Κατόπιν, 12% είναι εμπορία για την αφαίρεση οργάνων για την διάπραξη εγκληματικών δραστηριοτήτων κτλ. Τώρα, δεν θα υπερβάλλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο πολιτική, ένα νομικό πλαίσιο που δεν είναι μόνο πλήρη, αλλά επικεντρώνεται και στα θύματα. Η οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορία ανθρώπων ήταν ένα νέο μέσο, ήταν το πρώτο μέσο που υιοθετήθηκε υπό το ποινικό δίκαιο κατόπιν της υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας, αυτό το κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας. Η οδηγία αυτή δημιουργεί το πλαίσιο λοιπόν, πρόκειται για ένα μέσο το οποίο δίνει ένα κοινό ορισμό στο στο, έγκλημα, στο αδίκημα αυτό, επικεντρώνεται και στο φύλλο λαμβάνει υπόψη και τα παιδιά και επικεντρώνεται στα θύματα. Έχουμε μια μεγάλη σειρά διατάξεων για τα θύματα. Πρόσφατα το Δεκέμβριο δημοσιεύσαμε την πρώτη έκθεση της μεταφοράς της νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο. Ω θεματοφύλακα συνθήκης η Κομισιόν έλεγξε σε ποιο βαθμό έχουν μεταφέρει ορθώς ε, τα κράτη-μέλη την νομοθεσία στο εσωτερικό τους δίκαιο. Όλα τα κράτη-μέλη κοινοποίησαν ότι έχουν προβεί σε μεταφορά της νομοθεσίας. Ε, τώρα είμαστε σε διμερείς επαφές με τις κυβερνήσεις. Απλώς να σας πω ότι εξακολουθούμε να έχουμε εντοπίσει τομείς όπου χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες, παρόλο που και θέλω να τονίσω τις μεγάλες προσπάθειες που ήδη έχουν γίνει από τις 28 χώρες. Τώρα, οι τομείς όπου θέλουμε να γίνει περισσότερη δουλειά είναι συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τα παιδιά, πρέπει να δούμε περαιτέρω διατάξεις ε, σε ό,τι αφορά ε, το τεκμήριο της παιδικής ηλικίας, της παιδικής ηλικίας, την προστασία των θυμάτων ε, πριν και κατά τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών, αποζημίωση των θυμάτων, δηλαδή να μην τιμωρούνται τα θύματα λόγω για τα εγκλήματα που αναγκάστηκαν να διαπράξουν κατά τη διάρκεια της εμπορίας τους και μέτρα υποστήριξης της οικογένειας των θυμάτων το πολιτικό πλαίσιο στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της εμπορίας έρχεται σε ένα τέλος και τώρα αναπτύσσουμε το πλαίσιο για μετά το 2017. Όμως η εμπορία ανθρώπων σχετίζεται και με πολλές άλλες ε, πολιτικές, με πολλούς άλλους τομείς πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η στρατηγική ασφάλειας, η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, ε, η ευρωπαϊκή στρατηγική για το επιταναστευτικό κτλ. Επίσης, συζητήθηκε η εμπορία ανθρώπων και στην Σύνοδο της Βαλέτα, όπου τέθηκε ως προτεραιότητα και εργαζόμαστε ενεργά για το θέμα της εξωτερικής διάστασης. Συνεργαζόμαστε με τις μη ευρωπαϊκές χώρες για να οικοδομήσουν ικανότητες. Όπως ανέφερα νωρίτερα, Βλέπουμε τώρα ότι η εμπορία ανθρώπων ε, έχει κάνει τους ανθρώπους πιο ευάλωτους και το μεταναστευτικό πλαίσιο κάνει τους ανθρώπους πιο ευπαθείς ε, σε ε, δίκτυα εγκληματιών. Το γραφείο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος και των ναρκωτικών ανέφερε ότι πολλές από τις οδούς είναι ταυτόσιμες με αυτές τις μεταναστευτικές από τις οδούς, ε, τις εγκληματικές είναι ταυτόσιμες με τις οδούς της μετανάστευσης. Έχουμε δει ότι αυξάνεται το αριθμό των ασυνόδευτων ενηλίκων θα σας αναφέρω στατιστικά δεδομένα που έχουμε από την Ιταλία. Μας δείχνουν με σαφήνεια το επίπεδο του προβλήματος. Σύμφωνα με τον IOM και τη UNICEF για την περίοδο 2014-2015 η Ιταλία είδε αύξηση 300% στον αριθμό των θυμάτων από την Ιγυρία που φτάνουν στην Ιταλία και το ίμιση αυτών των ανθρώπων είναι ασυνόδευτα παιδιά. Στην περίπτωση της Ιταλίας με εκτιμά ότι το 80% των ε, γυναικών από την Ιγυρία που έχουν ταξιδέψει στην Ευρώπη είναι θύματα τράφικινγκ. Κυρίως για το σκοπό της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Βλέπουμε λοιπόν ένα νέο μια νέα τάση να φτάνουν τα θύματα του τράφικινγκ στι ακτέ Ευρώπη μέσω τη Λιβύη στην Ιταλία, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν και οδοί, χρησιμοποιούνται όλο ένα και περισσότερο τα αεροπλάνα, αλλά και η κεντρική οδός της Μεσογείου. Η εμπορία ανθρώπων ε, ουσιαστικά προκαλείται από μια σειρά παραγόντων, όπως είναι η ζήτηση και το κέρδος. Όμως ε, πολλά από αυτά δεν σχετίζονται με τη μετανάστευση αυτή καθ' αυτή. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι η απελπισία των ανθρώπων, των ε, μεταναστών, ε, των προσφύγων ε, μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση από τους διακινητές. Επίσης, τι ακόμα από τη Europol είναι ότι οι διακινητές Ουσιαστικά όλο και περισσότερο καταχρώνται τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών, συστήματα που αρχικά είχαν σχεδιαστεί για να ε, βοηθήσουν, να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους που φεύγουν από σειράξεις, ε, χρησιμοποιούνται όλο ένα και περισσότερο ε, για να νομοποιηθεί η διαμονή των ανθρώπων που είναι αντικείμενο τράφικινγκ και να μπορούν να μετακινηθούν στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, τα θύματα του τράφικινγκ ε, θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία στο σημερινό πλαίσιο της αναθεώρησης ε, του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασυλίου τα θύματα εμπορία ανθρώπων αναγνωρίζονται ω ειδική κατηγορία με ειδικέ ανάγκες. Και αυτό αντικατοπτρίζεται πολύ καλά στην ε, αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής, στην οδηγία για τα ελάχιστα, για τις ελάχιστες, μάλλον στην οδηγία, συγγνώμη, για τις διαδικασίες και στον κανονισμό του Βλήνου 3 όπου σύμφωνα με την πρόταση θα πρέπει να δοθεί δική έμφαση στα παιδιά κυρίως όταν ε, μιλάμε για τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού και την αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων. Τώρα, τι βλέπουμε εδώ. Ότι η εμπορία ανθρώπων μπορεί να συνδεθεί όντως με τα συστήματα ασύλου και το ΕΑΣΟ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για το Άσυλο, κοντεύει να ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο εργαλείο για το πώς θα μεταχειρίζεται τα θύματα του τράφικινγκ στο πλαίσιο διεθνών διαδικασιών. Αυτό είναι ένα εργαλείο σε δύο στάδια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εξ αποστάσεως, αλλά περιλαμβάνει και μια σειρά υλικών στοιχείων κατάρτισης. Υπάρχει και ένα εργαλείο κατάρτισης ε, στο διαδίκτυο και πάλι από το ΆΣΟ για να εντοπίζονται οι άνθρωποι που έχουν ειδικέ ανάγκες ε, και φυσικά εκεί περιλαμβάνεται και εμπορία ανθρώπων. Η Frontex έχει ουσιαστικά εκπονήσει μια σειρά προφίλ κινδύνου και μια σειρά εγχειριδίων για τους αξιωματούχους της που έχουν νόμιμη υποχρέωση να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και το νωρίτερο δυνατό να μπορούν να εντοπίσουν ένα ενδυνάμει θύμα εμπορίας. Όλες αυτές οι πληροφορίες διατίθεται στην ιστοσελίδα, στην Ευρωπαϊκή Ιστοσελίδα κατά του τράφικινγκ και είναι μια οριζόντια ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί έχουμε τη σχετική νομοθεσία, την ομολογία, τις διάφορες δημοσιεύσεις. Ε, μια άλλη εξέλιξη που θα λάβει η χώρα στο 2017 έχει να κάνει με το σύστημα πληροφοριών Schengen. Ακούμε ότι πολύ συχνά εξαφανίζονται παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε αυτά τα παιδιά. Και στο πλαίσιο της αναθεώρησης ε, του ΣΥΣ, θα συμπεριληφθεί ένα νέο εργαλείο στο σύστημα, όπου θα υπάρχει σαφής κατηγοριοποίηση Δηλαδή, όταν ε, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει εξαφανιστεί, μπορεί να υπάρχει παραπομπή σε κάποιο εξαφανισμένο παιδί και θα υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην εμπορία ανθρώπων. Αυτό θα γίνει το 2017. Όμως, επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά έρχονται πάρα πολύ αργά. Δηλαδή τα εργαλεία εντοπισμού, οι καταρτήσεις, οι μηχανισμοί κατάρτισης κτλ. έρχονται μετά τη χρηματοποίηση των ανθρώπων. Είναι πολύ αργά για αυτούς. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να επικεντρώσουμε τώρα τις προσπαθίες μας στην πρόληψη. Ξέρουμε και θέλω να πιστήσω την προσοχή σας στο εξή ότι η εμπορία ανθρώπων είναι μία μορφή εγκλήματος, ιδιαίτερα κερδοφόρος. Δεν υπερβάλλουμε να λέμε ότι ουσιαστικά ένας πόλος έλξης είναι η ζήτηση, αλλά ουσιαστικά κινητοποιείται και λόγω του κέρδους. Η Europol εκτιμά ότι 29,4 δισεκατομμύρια είναι το παγκόσμιο ετήσιο προϊόν. Με 23,4 δις να είναι μόνο το κέρδος της εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση. Σκεφτείτε εδώ τους αριθμούς. Είναι σημαντικό, γιατί αν είμαστε εδώ για την πρόληψη, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι στοχεύουμε στα κέρδη αυτά και θα κάνουμε αυτό το έγκλημα υψηλού κινδύνου, δηλαδή θα επιτεθούμε στους διακινητές εκεί όπου τους ενδιαφέρει περισσότερο στο κέρδος και η εμπορία γεννά κέρδος όχι μόνο για τους διακινητές, αλλά φέρνει κέρδος και για νόμιμους τομείς, αλλά και παράνομους τομείς της οικονομίας μας. Μπορούμε να έχουμε όχι μόνο το παράνομο τομέα, αλλά μπορούμε να έχουμε και νόμιμες επιχειρήσεις που να εμπλέκονται κατά κάποιο τρόπο. Σκεφτείτε τις αλυσίδες ε, εφοδιασμού. Σκεφτείτε τη μεμονωμένη μας ευθύνη ως καταναλωτές και εδώ θέλω να τονίσω ότι η οδηγία κατά του τράφικιν έχει ένα μέρος για την πρόληψη. Υποχρεώνει νομικά τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι μειώνεται η ζήτηση. Εκεί επικεντρώθηκε η πρώτη έκθεση πρόοδου που σας ανέφερα πριν. Βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη μας ανέφεραν ότι έχουν κάνει μία σειρά διαδικασιών κατάρτισης για να ταυτοποιούνται τα θύματα δεόντας, όμως ε, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η σύνδεση με την πρόληψη. Εμείς ε, είδαμε μέτρα τα οποία ουσιαστικά θεωρείται ότι ποινικοποιούν αυτούς που χρησιμοποιούν ε, αυτό το δίκτυο. Σκεφτείτε, παραδείγματος χάρη, άλλες περιπτώσεις, κάποιο έγκλημα που Παραδείγματο χάρη το άτομο το οποίο χρησιμοποιεί τι υπηρεσίε ε, δεν αντιμετωπίζει τον νόμο. Ε, η Κομισιόν ε, παρουσίασε την έκθεσή μας στο Κοινοβούλιο σε σχέση με τα δίκτυα ε, που, ανθρώπων που χρησιμοποιούν ουσιαστικά αυτές τις υπηρεσίες. Μόνο 10 κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι ποινικό αδίκημα η χρήση των υπηρεσιών των βήματων του τράφικινγκ για όλες τις μορφές εκμετάλλευσης. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί, τι βλέπουμε. Ότι υπάρχει διαφορετική νομική μεταχείριση. Κάτι που δεν μας βοηθά στην πρόληψη του εγκλήματος. Σε αυτό το περιβάλλον των ε, διάφορων νομικών πρακτικών ανθεί το έγκλημα. Ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα επιδέξη οι διακινητές ε, στο να μπορούν να εκμεταλλευτούν κάποια κενά ή διαφορές στην νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι είδαμε. Ότι ουσιαστικά ε, αυτό έχει παρενέργειες στο έγκλημα. Αν δεν έχουμε όμως μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διασφαλίσουμε ότι όσοι χρησιμοποιούν ε, τα θύματα ποινικοποιούνται, τότε τι κάνουμε εδώ, διατηρούμε έναν πολιτισμό ατιμορρησίας. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Έχουμε διανύμει την έκθεση στους συναδέλφου στα κοινοβούλια. Είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα μας. Αναφέρει διάφορα μέτρα και προσεγγίσεις, αλλά τι λέμε εμείς. Ότι είναι ζωτική σημασίας και επίγει να δούμε τα στοιχεία της πρόληψης, να δούμε το γεγονός ότι εδώ μιλάμε για ζήτηση και ότι το τράφικινγκ αφορά πέρα από τη ζήτηση και το κέρδος. Αυτό που θεωρούμε σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τα θύματα του τράφικινγκ τα αντιμετωπίζουμε ως ανθρώπους με δικαιώματα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαιώματα, δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα αυτά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όσοι εκμεταλλεύονται τα τροτά σημεία των ανθρώπων, το γεγονό ότι βρίσκονται σε διάφορες καταστάσεις και τις μεταναστευτικές ε, τους, σχέδια, θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Και υπάρχει μια βούληση να γίνουν περισσότερα. Αν υπάρχει αυτή η βούληση, τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος. Θα σταματήσω εδώ, θα απαντήσω σε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Ευχαρίστω, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, να σας απαντήσω. Thank you ε, Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβασή σας. Ε, νομίζω ότι έχουμε στη διάθεσή μας αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε και για να μπορέσουμε να θέσουμε ερωτήσει. Και ας αρχίσουμε με τον κύριο Γιώργιο Πάλι από την Ελλάδα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καταρχήν θα σας πω εξ αρχής ότι οι περιορισμοί, εξειδικεύσεις και τελικά οι αποκλεισμοί νομοτελειακά αποτελούν ε, την πηγή του άλλου δρόμου, την πηγή της παράνομης κίνησης των ανθρώπων. Το τράφικινγκ. Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ του 2015, όπως το βίωσα εγώ στη Λέσβο, τη βασική πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη, και της περίοδου μετά την αντιευρωπαϊκή πολιτική των χωρών του Βίζεγκραντ και κατ' επέκταση και την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ε, μας, μας δείχνει χαρακτηριστικά του τι συνέβη. Το 2015 η Ελλάδα αποτελούσε μια όαση για τους πρόσφυγες, για τους πρόσφυγες κυρίως. Ε, ήταν εφικτή η ελεύθερη κίνηση των ανθρώπων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μετά την καταγραφή τους μεταφέρονταν από τα νησιά του Αιγαίου στην υπηρετική Ελλάδα και από εκεί ακολουθούσε έναν νόμιμο τρόπο με τα αντίτιμα που αποτελούν ε, τη μετακίνηση του όπως ο κάθε άνθρωπος. Αυτό αφαιρούσε ουσιαστικά το οικονομικό αντικείμενο στους διακινητές. Είχαμε την απεμπλοκή από τα δίκτυα των διακινητών και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στην πορεία αυτή ε, απαλλάχθηκαν από αυτόν τον φαύλο κύκλο της, ε, του τράφικινγκ. Ε, από εκεί και πέρα όμως έχουμε τον εγκλωβισμό των ανθρώπων. Είναι κάτι που το βιώνουμε και τώρα. Οι εγκλωβισμένοι άνθρωποι αναγκάζονται να αναζητήσουν άλλες οδούς για να ξεφύγουν ε, καταρχήν από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που είναι εγκλωβισμένοι μέσα στην ίδια τη χώρα την Ελλάδα, σε, με εσωτερικά σύνορα. Τα θύματα που έχουμε είναι θύματα πρόσφυγες και μετανάστες θύματα του τράφικινγκ, αλλά έχουμε και μια έξαρση πια ε, των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Το νομικό πλαίσιο έχει γίνει σκληρό. Με καλά και κακά αποτελέσματα. Ένα από τα κακά αποτελέσματα είναι ότι στις ελληνικές φυλακές βρίσκονται δεκάδες άνθρωποι με πολιτής καθήρξης, ε, με την κατηγορία των διακινητών. Θα σας αναφέρω μόνο ότι το 50% των, των κρατούμενων στις φυλακές ανηλίκων στην Ελλάδα είναι ξένοι ε, κρατούμενοι οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί με πολιτικές καθήξεις ως διακινητές. Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Ε, το ελληνικό κράτος έχει κάνει μεγάλο αριθμό ενεργειών ούτως ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Ε, δεν θα μπορέσει να γίνει κάτι αν δεν καταλάβουμε όλοι μας ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το τράφικ είναι να αφαιρέσουμε το οικονομικό αντικείμενο που είναι οι περιορισμοί που βάζουμε στους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Yes, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Γιούχο Έρχολα. Ελπίζω να είπα σωστά το όνομά του. Εάν δεν το είπα καλά, λοιπόν, πολύ. Ορίστε, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλή ήταν η προφορά σας. Αρκετά ευκρινές το όνομά μου. Το κλειδί για να αντιμετωπιστεί το θέμα είναι να δίνονται πληροφορίες, ενημέρωση στους ανθρώπους εκεί όπου, όπου είναι η αφετηρία και όπου ξεκινούν. 12 χρόνια έχω δουλέψει με ανθρώπους που ζητούν άσυλο. Και έχω διαπιστώσει ότι πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς δεν είναι πραγματικοί πρόσφυγες, αλλά μετακινούνται για οικονομικούς λόγους. Και επειδή το επίπεδο των προσόντων τους είναι συνήθως πολύ χαμηλό, δεν έχουμε την δυνατότητα να τους προσλάβουμε, να τους ε, ε, δώσουμε δουλειές. Αποτελούν τελικώς οικονομική επιβάρυνση. Πολλοί από αυτούς που ζητούν άσυλο ε, έχουν και μεγάλα χρέη, χρωστούν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στους διάφορους διακινητές και επειδή δεν υπάρχουν αρκετές δουλειές τελικώς πέφτουν είτε στην ε, γκρίζα λεγόμενη οικονομία είτε στην εγκληματικότητα. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου η Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι μαζί να αρχίσουμε μια μαζική προσπάθεια ενημέρωσης των ανθρώπων στους τόπους προέλευσής τους ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην ξεκινούν καν το ταξίδι προς την Ευρώπη. Να ενημερωθούν για όλους αυτούς τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Σκλαβιά, ε, σεξουαλική εκμετάλλευση, το ίδιο το ταξίδι όταν ξεκινούν οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν πού θα καταλήξουν. Είναι θύματα των διακινητών οι οποίοι τους γεμίζουν ψέματα. Τους λένε ότι «Α, κοιτάξτε, σας περιμένουν καλές δουλειές, με καλές συνθήκες, στην Ευρώπη σας περιμένουν ανοιχτές αγκαλιές». Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν θύματα και ο μόνος τρόπος για να τους βοηθήσουμε, ξαναλέω, είναι μια μαζική προσπάθεια ενημέρωσης στις χώρες τους. Η πρόταση. Έχει καλώ. Τώρα, ο Λόρδος Σόλε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ σημαντικό θέμα και ασφαλώς η αστυνόμευση θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Επανέρχομαι στο θέμα των ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών. Εμείς της Βουλής των Λόρδων έχουμε συντάξει μια έκθεση που μπορείτε να την βρείτε κιόλας για τα ασυνόδευτα παιδιά για τους ασυνόδευτους ε, νεαρούς μετανάστες δηλαδή. Όταν συλλέξαμε ε, ε, ενδείξει και στοιχεία από διάφορα πρόσωπα, είδαμε ότι ένα ασυνόδευτο παιδί, εφόσον του βρεθεί από την αρχή ένας κηδεμόνας, από την αρχή της έλευσής του, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να πέσει σε ε, μεγάλους κινδύνους. Στην περίπτωσή μας έχουν χαθεί δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Στην περίπτωση που συζητούμε δεν γνωρίζουμε που έχουν καταλήξει. Είτε τους βάζουν σε κάποιες δουλειές τύπου σκλαβοπάζαρου, είτε για σεξουαλικές ε, για σεξουαλική εκμετάλλευση. Έχω μιλήσει μάλιστα και με ένα Γερμανό δικαστή και μου είπαν ότι έχουν ένα σύστημα και μόνον. Εφόσον υπάρχει ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, διορισμένο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προστασία και ευημερία του παιδιού, έχουμε τουλάχιστον έναν τρόπο να προστατεύσουμε το παιδί σε, από αυτό το τρομερό εμπόριο. Ευχαριστώ. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να αντιμετωπιστούν και όλες αυτές οι συμμόριες. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Πάλι. Μήπως μπορείτε να επαναλάβετε, μήπως μπορείτε να συνοψίσετε πάλι την ομιλία σας. Γιατί η μετάφραση δεν ήταν ε, σωστή. Η μεταφορά το διάστημα του 2015 γινόταν με την νόμιμη οδό, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς με το ίδιο αντίκτυπο όπως σε όλους τους πολίτες, είτε ήταν ε, πρόσφυγες και μετανάστες, είτε πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δεν είχε οικονομική επίπτωση, ήταν κάτι θετικό, ήταν μικρό το κόστος της μεταφοράς των ανθρώπων, γιατί πληρώνουν το εισιτήριο όπως πληρώνουν κάθε πολίτης. Ε, και μια διευκρίνηση ακόμα ότι η λύση για να αφαιρέσουμε το οικονομικό αντικείμενο από τους διακινητές είναι η νόμιμη οδός μετακίνηση των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ. Νομίζω ήταν πράγματι χρήσιμο που επαναλάβατε. Η κυρία Οντέκη Λόνε από την Εστονία. Όντως, το ε, λαθρεμπόριο ανθρώπων προκαλείται από τη, ζήτηση, ε, από τη ζήτηση. Ε, Βεβαίω και πρόκειται και για την ε, γενετήσια κατάχρηση και ούτω καθεξής. Ε, υπάρχουν και κάποιες νόμιμες πτυχές. Οι περισσότεροι οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι συνήθως ακολουθούν τις ίδιες οδούς και μπαίνουν από τις ίδιες εισόδους όπως οι ετούντες άσυλο, πολλοί από αυτούς πέφτουν θύματα εγκληματικών δικτύων. Βρίσκουν όμως δουλειές είτε στη γεωργία μας, είτε στη βιομηχανία. Φτιάχνουν, ε, ε, παράγουν ρουχισμό ή κάνουν ακόμα και μανικιούρ σε ανθρώπους που μερικοί από αυτούς μπορεί να βρίσκονται και μέσα στην αίθουσα. Άρα λοιπόν αυτό το ε, εμπόριο ανθρώπων θα είναι επικερδές μέχρι ότου πείσουμε εμείς τον κόσμο ότι να αντιληφθούμε ότι δεν είμαστε διατηθειμένοι να το δεχτούμε αυτό και δεν θα τους πληρώνουμε λιγότερα για να κάνουν τις βρώμικες δουλειές στους ανθρώπους αυτούς. Αντί να υποσχόμεθα ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, στην ουσία έχουμε φτιάξει ένα σύστημα ελεύθερης διακίνησης μισθών και αμοιβών και οι λαθρέοι διακινητές το εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα για να σταματήσει αυτή η φοβερή κατάσταση μέσα σε αυτά τα κλιματικά δίκτυα που παγιδεύονται οι άνθρωποι, πρέπει να δράσουμε με τρόπο οικονομικό. Πρέπει δηλαδή να ρίξουμε το βάρο μα στου μισθού, στα μισθολογικά των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη, στι συνθήκε εργασία, Για να πάψει αυτό το λαθρεμπόριο ψυχών σημαίνει ότι πρέπει να καταστρέψουμε την ζήτηση. Την ζήτηση για τη σκλαβιά, για του ανθρώπου που δουλεύουν υπό συνθήκες σκλαβιά. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα... Φρανκ Τρούτσεκ, Σλοβενία. Μπορώ να τα πω στα σλοβενικά, λέει ο κ. Τρούτσεκ. ναι. Όπως είπε προηγουμένως μια συνάδελφός μου από ε, βαλτική χώρα, είπε κάτι σωστό δηλαδή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει κοινωνική ένωση και τότε μόνο θα παραμείνει ενωμένη γιατί αλλιώς θα διαλυθεί. Είναι γεγονό ότι μιλούμε για εκμετάλλευση από εγκληματικά δίκτυα, πρόκειται δηλαδή για business και φτάνουν στο, στα τρία τέταρτα του εθνικού προϊόντος της ε, Σλοβενίας. τα είπε και αμέσω προλαλήσασα, ότι τελικώ οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν υπό συνθήκε σκλαβιά για να παράγουν εμπορεύματα. Η Σλοβενία είναι μικρή χώρα, αλλά έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα ότι το θέμα αυτό είναι σαν περιβαλλοντικό, δηλαδή δεν γνωρίζει σύνορα, ξεπερνά τα σύνορα. Η Σλοβενία έχει περιορισμένους πόρους. Η Σλοβενία στην Σλοβενία μάλλον, όπως και σε ορισμένες παραμεθόριες χώρες, οι μη κρατικέ οργανώσεις έχουν περισσότερη γνώση του θέματος από τις ε, κρατικές αρχές. Ο συνάδελφός μας από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης μας έδωσε ένα παράδειγμα από την πράξη σχετικά με αυτό το σύστημα κηδεμόνων. Όταν μιλούμε για λαθρεμπόριο ανθρώπων, αν θέλουμε να σπάσουμε τον φαυλοκύκλο πρέπει να, σπάσει, να σπάσουν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας. Δηλαδή, θα συγκρουστούμε και με κάποιες πολιτιστικές πρακτικές που δεν είναι πια αποδεχτές. Για παράδειγμα, ε, η μοίρα των ανηλίκων στις κοινότητες Ρωμά. Πρόκειται για μια πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τρόπο συνολικό. Και οι πολιτικοί πρέπει να διδαχθούν πολλά από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ωραία, εδώ ολοκληρώθηκε ο κατάλογος και μπορώ να ρωτήσω ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο τώρα, γιατί έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας μπορείτε να αντιρωτήσετε ό,τι θέλετε, πολλά πράγματα. Ε, γιατί αυτή είναι μια ευκαιρία για τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μια ευκαιρία που τους δίνεται. Ενδιαφέρεται κανείς άλλος? Okay, then I... Ωραία. Εάν όχι, εγώ θα κάνω κάποιες ερωτήσεις ε, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς, τι γίνεται με τα κράτη-μέλη. Πώς ε, αντιμετωπίζουν ε, την οδηγία αντι-trafficking τα κράτη-μέλη. Ε, δηλαδή η, εφαρμογή γίνεται σωστά, τα πράγματα πάνε καλά ή σε ποιες χώρες χρειάζεται μια όθηση, πρέπει να είναι πιο πετυχημένη δηλαδή η εφαρμογή. Και μετά στην Ευρώπη οι, ε, οι αγοραπολισίες οργάνων, το εμπόριο οργάνων. Πώς είναι σημαντικό στην Ευρώπη, έχουμε την περίπτωση του κοσυφοπεδίου. Στην μελέτη σας ε, έχετε αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Και όπως είπε και ένας προηγούμενος ομιλητής, η εκμετάλλευση της εργασίας είναι σημαντική και αυτή είναι μεγάλο το ποσοστό δηλαδή. Αυτά είναι τα τρία ερωτήματά μου. Άλλες ερωτήσεις. Μετά το κλείσιμο των συνόρων ε, στη Βαλκανική, αν υπάρχει μετρήσιμο και σε ποιο ποσοστό υπάρχει, αν υπάρχει αύξηση ε, της καταγραφής του τράφικινγκ ε, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Any other questions? Άλλες ερωτήσεις ή συνεισφορές ενδεχόμενα, παρεμβάσεις, όπως θέλετε πέστε τις. Ωραία. Εάν όχι, έχετε το λόγο. Σας δίνω το λόγο ξανά, κυρία Σακελιάδου, και έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε πλήρως. Λοιπόν, μου δίδεται την ευκαιρία να επανέλθω σε κάποια θέματα που αφορούν τα τελευταία μας ευρήματα. Και θα ξεκινήσω με τις τελευταίες τάσεις. Η Κομισιό το Μάιο του 2016 δημοσίευσε την πρώτη έκθεση πρόοδου, όπου ακριβώς κατέγραφε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην καταπολέμηση της ε, ε μετακίνησης των ατόμων. Και ε, είδαμε ότι διαμορφώνονται κάποιες νέες τάσεις. Δηλαδή, τι εννοώ. Έχουμε μία αύξηση στην διακίνηση των παιδιών, των ανηλίκων. Τα παιδιά ούτως ή άλλως ε, φαίνεται ότι πέφτουν στην παγίδα αυτής της ε, διακίνησης και η διακίνηση γίνεται επίσης και ε, μέσα στα πλαίσια αναγκαστικών ή ψεύτικων γάμων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε θύματα εκμετάλλευσης, ε, θύματα τα οποία έχουν ε, προβλήματα ψυχολογικά, τα θύματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ένα άλλο, μια άλλη τάση που βλέπουμε μέσα στα πλαίσια της ε, παράνομης διακίνησης ε, για λόγους ε, αναγκαστικής εργασίας είναι ότι οι γυναίκες πέφτουν θύματα κυρίως και Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι δύσκολο να επιληθεί από ό,τι μας λένε. Επίσης είναι ένας τομέας ακριβώς ο οποίος έχει σαν στόχο κυρίως τις γυναίκες. A Ένας, μια σειρά τομέων έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, όπως η γεωργία, ε, οι οικοδομές, ε, ξενοδοχεία εστιατόρια. Αυτοί είναι οικονομικές δραστηριότητες, αυτές είναι οι οικονομικές δραστηριότητες όπου υπάρχουν ε, άτομα τα οποία είναι θύματα παράνομης διακίνησης. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ε, ασφαλής από την ε, παράνομη διακίνηση. Όλοι, όλους μας αφορά και όλοι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε να δώσουμε μία απάντηση ε, σφαιρική και αποτελεσματική στο πρόβλημα αυτό. Τα κράτη-μέλη έχουν μεταθέσει στην εθνική του νομοθεσία την οδηγία. Άρα μια υποχρέωση έχει υλοποιηθεί. Και αυτό είναι το αντικείμενο το οποίο ε, ήταν, ήταν το αντικείμενο της έκθεσης της οποίας δημοσιεύσαμε το Δεκέμβριο του 2016. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα, πολύ περισσότερα, ε, ε, υιοθετώντας διατάξεις ε, που να αφορούν αποκλειστικά τα θέματα προστασίας των ανηλίκων. Είναι και θέματα κυδαιμονίας, παραδείγματο χάρη. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δημιουργεί υποχρεώσεις στα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν τα παιδιά ορίζοντας κυδαιμόνες. Επίσης είδαμε ότι οι διατάξεις δεν ήταν πολύ σαφές όσον αφορά την έννοια της της παιδικής ηλικίας, του παιδιού. Δηλαδή, εάν τα, οι αρχές θεωρούν ότι το άτομο το οποίο έχουν μπροστά τους έχει σοβαρές πιθανότητες να είναι παιδί, να είναι ανήλικας, πρέπει να τα αντιμετωπίσουν έτσι, ως παιδί, ως ανήλικα. Επίσης δεν υπάρχουν διατάξεις όσον αφορά την αποζημίωση των θυμάτων, διότι έχουν δικαίωμα σε αποζημίωση, έχουν δικαίωμα να εισπράξουν κάποια χρήματα. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε και την έννοια της μη τιμω, τιμωρίας των θυμάτων. Ας πούμε, η διακίνηση γίνεται πολλές φορές και για κλιματικές δραστηριότητες. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι τα θύματα διακίνησης χρησιμοποιούνται πολλές φορές από τους εγκληματίε για να ε, εκτελέσουν κάποιες εγκληματικές δραστηριότητες, να γίνουν βαποράκια, να ε, ε, κλέψουν ένα, σπίτι. Αυτά όμως είναι θύματα, δεν πρέπει να είναι αυτά τα οποία θα βρεθούν πίσω τα κάγκελα. Πρέπει να τιμωρήσουμε τους δράστες τους αυτούργους. Επίσης, πρέπει να βοηθήσουμε τις οικογένειες των θυμάτων ε, της διακίνησης. Επιτρέψτε μου να μην πω σε λεπτομέρειες που αφορούν συγκεκριμένες χώρες, γιατί δεν είναι το αντικείμενο της έκθεσης αυτό. Ε, εδώ προσπαθούμε να ερευνήσουμε τα πορίσματα ε, της έκθεσης ε, της μεταφοράς της ε, κοινοτικής οδηγίας στην Εθνική Νομοθεσία και εάν όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσε ότι δεν έχει γίνει σωστά η μεταφορά αυτή, θα το εξετάσουμε. Όμως αυτή τη στιγμή εξετάζουμε αυτή την ε, εθνική νομοθεσία, αλλά και την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Με ρωτήσατε για, την, ε, το λαθρεμπόριο οργάνων. Όντως είναι μια μορφή εμπορίου που ανθεί. Δεν έχουμε βέβαια στατιστικά στοιχεία αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να τονίσω βέβαια ότι σας δίνω στατιστικά στοιχεία. Δεν σας δίνω, δεν σας παρουσιάζω εκτιμήσεις ή ε, φουσκωμένα νούμερα. Όχι. Μιλάω για, με στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να καταγράψουν και να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Και εδώ τίθεται ένα θέμα που έθεσε και ο ε, βουλευτής από την Ελλάδα, ότι τα δεδομένα τα οποία έχουμε δεν παρουσιάζουν πλήρως την ε, εικόνα στην Ευρώπη. Ακούμε ότι στην, ε, η κατάσταση των, στα σύνορα έχει επιδεινώσει την, ε, την εικόνα της διακίνησης και ιδίως τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα. Όμως αυτή την κατάσταση, αυτή την εικόνα δεν μπορούμε να την μεταφράσουμε σε στατιστικά στοιχεία. Εγώ θεωρώ ότι όντως τα νούμερα είναι σημαντικά. Πρέπει να χρησιμοποιούμε νούμερα για να βελτιώσουμε τις πολιτικές μας. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστούμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουμε το σύστημα συλλογής των ε, ε, δεδομένων. Όμως... <clears throat> Πρέπει να έχουμε ε, αδιάσυστα αν θέλετε στοιχεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ε, η διακίνηση για την αφαίρεση οργάνων, δηλαδή διακίνηση ανθρώπων, η διακίνηση των ανθρώπων για την αφαίρεση οργάνων είναι διαφορετικό από την διακίνηση των οργάνων. Υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχουμε διάφορα project και θα έχουμε χρηματοδοτήσει και project. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να έχουμε στο μέλλον στοιχεία που θα αφορούν και τα δύο ε, και τους δύο τομείς. Ένα άλλο τομέα είναι η διακίνηση για παράνομες υιοθεσίε, για την πώληση των παιδιών. Εδώ εντάσσονται μεγάλες κατηγορίες, όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και ε, διάφοροι επαγγελματίε συμμετέχουν ε, σε αυτή τη διακίνηση. Όταν μιλάμε για διακίνηση ανθρώπων για, το, για την αφαίρεση οργάνων, φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει κανείς εάν δεν συμμετείχαν στο κύκλωμα και γιατροί, ας πούμε. Και αυτό αναφέρθηκε προηγουμένω ότι θα, θα πρέπει να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση. Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση πολυτομεακή, αν θέλετε. Ε, διότι η διακίνηση των ανθρώπων δεν είναι μόνο θέμα αστυνομικό, είναι θέμα της αστυνομίας βέβαια, είναι θέμα της κοινωνικής πολιτικής, της προστασίας των συνόρων, της ε, ε, παιδείας, θέμα που αφορά τους γιατρούς και το προσωπικό, το ιατρικό. Δηλαδή είναι θέματα, θέματα τα οποία άπτονται όλων των ε, κοινωνικών ε, στρωμάτων, ε, τάξεων, κατηγοριών. Δηλαδή, και θα πρέπει αυτοί οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα θύματα της διακίνησης πρέπει να ξέρουν να είναι εκπαιδευμένοι και να ξέρουν αυτό το οποίο ονομάζουμε δίκτυ διακίνησης. Θα έχετε ακούσει πολλέ φορέ τον συντονιστή να λέει ότι κοιτάξτε γύρω σας, θα δείτε σίγουρα θύματα διακίνησης ε, ε, στο δρόμο να περπατάνε δίπλα σας. Τι λέμε. Εμείς λέμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο το οποίο δίνει κάποια δικαιώματα ε, στους, στα θύματα, υποστήριξης, βοήθειας κτλ. Όμως, εάν δεν αναγνωριστούν τα άτομα αυτά ως θύματα διακίνησης, ε, δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε και αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν έχουμε μαζικές αφήξεις δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουμε να ε, εξασφαλίσουμε οι υπεύθυνοι να, περνάνε, να περάσουν αρκετό χρόνο με, τα, με, τα, με τους μετανάστες για να μπορέσουν να εφαρμοστούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και επομένως να είναι ε, εύκολα θύματα της διακίνησης. Στην αρχή του 2015 δημοσιεύσαμε μία έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, την, για τον αντοπισμό των θυμάτων ανθρώπινης διακίνησης στην διαδικασία ασύλου. Το κάναμε αυτό και είδαμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών κατάλαβαν ότι μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι ανάμεσα στην, στην όλη διαδικασία για την χορήγηση ασύλου και στην παράνομη διακίνηση. Όμως πολλές φορές ε, οι ίδιοι που ζητάνε άσυλο δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το σύστημα χορήγησης ασύλου και αυτό δημιουργεί προβλήματα και στην διοικητική αρχή που είναι υπεύθυνη τη χορήγηση του ασύλου, αλλά και στα θύματα αυτά καθεαυτά, διότι τα θύματα τελικά, τα άτομα αυτά μάλλον, οι υποψήφοι αυτοί, ε, γίνονται ευάλωτοι και ανοιχτοί σε συνεκμετάλλευση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχουν περάσει τα άτομα αυτά. Όχι μόνο όταν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δούμε και τι τραβήξανε πριν περάσουν ε, στις ακτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία το 65% των καταγεγραμμένων θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι τα θύματα της διακίνησης δεν μας έρχονται μόνο απ' έξω, αλλά είναι και μέλη της δικής μας οικογένειας. Ε, προέρχονται από τα δικά μας κράτη-μέλη. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε η διακίνηση ήταν παρούσα και πριν την μεταναστευτική κρίση και τώρα και μετά. Απλώς έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση τα... υπάρχουν πολύ περισσότερα θύματα ευάλωτα ε, στην διακίνηση είναι πολύ πιο εύκολα να πέσουν στην παγίδα των διακινητών ε, τα άτομα αυτά. Και ε, ε, θα πρέπει να έχουμε σαφείς έννοιες. Το λέει και ο συντονιστής. Άλλο είναι η διακίνηση και άλλο είναι η παράνομη είσοδος, αυτοί που βοηθούν την παράνομη είσοδο. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Τώρα, αυτοί οι οποίοι βοηθήθηκαν να, εισά, να, να, να μπουν ε, ε, παράνομα ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς δεν μας ε, αποκλείει το γεγονός ότι μπορούν όντως μετά να είναι θύματα της παράνομης διακίνησης. Αλλά Όταν μιλάμε για παράνομη διακίνηση, δεν μιλάμε μόνο για διέλευση συνόδων, συνόδων, συνόρων. Ε, συνεχίζει το έγκλημα, αν θέλετε. Γι' αυτό θα πρέπει να μπορούμε να προστατεύσουμε τα άτομα τα οποία χρειάζονται προστασία. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ε, στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να, να προσέξουμε επομένως όταν χρησιμοποιούμε διάφορες, ε, ε διάφορους όρους ότι το trafficking δεν είναι το ίδιο με το smuggling, δηλαδή η διακίνηση δεν είναι το ίδιο με την παράνομη είσοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και για τη τελευταία παρατηρήσή σας. Τι είναι δηλαδή η εμπορία ανθρώπων και τι δεν είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αποφάσει που λαμβάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ότι λοιπόν, υπάρχει μια ερώτηση, παρακαλώ. Μια διευκρίνηση. Νόμιζα ότι είπατε ότι απέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις χώρες να υπάρχει μια διευθέτηση επιτροπίας σε κάθε χώρα. Νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. μπορείτε να διευκρινίσετε ή δεν σας άκουσα καλά. Ναι, η οδηγία αντιτράφικινγκ προβλέπει νομική υποχρέωση στα κράτη-μέλη να διορίσουν επίτροπο ή νομικό εκπρόσωπο των παιδιών που είναι θύματα τράφικινγκ. Να σας πω ότι πρόκειται για μια οδηγία που αφορά την εμπορία ανθρώπων. Τα παιδιά που δεν είναι θύματα τράφικινγκ δεν εμπίπτουν στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής. Υπάρχουν ε, άλλα νομοθετήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν διατάξει την Επιτροπή, όμως στην οδηγία αυτή για κατά του τράφικινγκ υπήρχε συγκεκριμένη διάταξη για τα παιδιά που είναι θύματα τράφικινγκ. Έχουμε δημοσιεύσει και ένα εγχειρίδιο σε συνεργασία με τον Οργανισμό Σεβασμού των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και παρέχουμε αρχές και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο να θεσπιστούν εθνικά συστήματα επιτροπίας για τα θύματα του τράφικινγκ, που μπορούν όμως να προσφέρουν υπηρεσίες και σε άλλα παιδιά. Μπορεί να υπάρχουν και σε άλλες διαδικασίες. Ελπίζω να σας ε, απάντησα. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Όμως, αν ε, κάνουμε κάτι τέτοιο για τα παιδιά που είναι θύματα τράφικινγκ, τότε φαίνεται να είναι ένα μικρό βήμα, ίσως να είναι ακριβό για κάποιες χώρες, αλλά μικρό βήμα για να πούμε ότι όλοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα έπρεπε να έχουν ένα επίτροπο. Πρέπει να διοριστεί ένας επίτροπος για αυτούς. Και στην έκθεση αυτή που έχουμε παράξει, το λέμε γιατί ξέρουμε ότι τουλάχιστον 10.000 παιδιά έχουν εξαφανιστεί και υπάρχουν και άλλε περιπτώσει τι οποίε δεν γνωρίζουμε. Πρέπει να υπάρχει τεράστιο αριθμό ανθρώπων, παιδιών που έχουν εξαφανιστεί. Ενώ αν έχει διοριστεί ένα άνθρωπος που είναι υπεύθυνο που ξέρει τι συμβαίνει και που είναι το παιδί και εκπροσωπεί αυτό το παιδί στις αρχές, τότε έχεις ένα πολύ καλύτερο τρόπο να σταματήσεις ε, τις εξαφανίσει. Και ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου ότι πολλές χιλιάδες των εξαφανισμένων ε, τελικά έχουν καταλήξει θύματα εμπορίας. Αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι εγώ μιλάω από μια συγκεκριμένη σκοπιά. Μιλώ εκ μέρου ε, τη συντρονή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη εμπειρία ανθρώπων. Και μιλάμε για παιδιά που είναι θύματα τράφικινγκ, είτε είναι ασυνόδευτα είτε όχι. Φυσικά όταν μιλάμε για γενικά πρότυπα σε σχέση με τα παιδιά, η Κομισιόν επίση έχει δεσμευτεί να προωθήσει το σεβασμό των διεθνών προτύπων του CRC και εργαζόμαστε προς την εκπόνηση μιας ανακοίνωσης που θα θίξει το θέμα της προστασίας όλων των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης και πιστεύω ότι η Επιτροπή είναι ένα από τα θέματα που θα περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση αυτή. Ξέρω ότι τα παιδιά που ήταν στο πλαίσιο του συστήματος ασύλου Υπάρχουν ε, και κάποιες ε, διατάξεις που σχετίζονται με την Επιτροπή στις διατάξεις που αφορούν το άσυλο, όμως ε, μπορεί να είναι κοινός να προσφέρει περισσότερη καθοδίκηση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το εγχειρίδιο που εκπονήσαμε σίγουρα μπορεί να καλύψει πολλές άλλες κατηγορίες παιδιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα. Όχι μόνο για τα θύματα εμπορίας. Αυτή ήταν η λογική όταν το εκπονήσαμε. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες, τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ε, είναι και προσβάσιμο σε εθνικό επίπεδο και μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα, στην Ευρωπαϊκή Ιστοσελίδα κατά του τράφικινγκ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, θα το έχω κατά νου. Απλώς να πω, αν 10.000 παιδιά έχουν εξαφανιστεί, είναι σχεδόν ε, αδύνατο να πιστέψουμε ε, ουσιαστικά ότι δεν είναι και θύματα τράφικινγκ. Επομένω, είναι ένα θέμα και νομοθεσία που αφορά το τράφικινγκ. Γι' αυτό στο σύστημα πληροφοριών ΣΕΝΚΕΝ ε, τώρα θα αναπτύξουμε αυτό το επιχειρησιακό εργαλείο όπου οι αρχές μπορούν να καταχωρήσουν πληροφορίες, μπορούν να ε, καταχωρήσουν ε, την πληροφορία ότι λείπει αυτό το παιδί, έχει εξαφανιστεί, είναι ασυνόδευτο ή είναι σε κίνδυνο να γίνει θύμα εμπορία. Έτσι λοιπόν, ελπίζουμε ότι τα επόμενα έτη θα έχουμε και σχετικά δεδομένα. Μάλιστα, είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Ορισμένα από τα εξαφανισμένα παιδιά, από τα γνώμενα παιδιά, πήγαν σε κάποια άλλη χώρα. Δεν ξέρουμε τώρα που βρίσκονται. Μπορεί να είναι με τις οικογένειές τους ή έχουμε μεγάλα προβλήματα με την εμπορία ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση. Δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε που είναι οι άνθρωποι, αν είναι θύματα ή όχι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για τα παιδιά. Χρειάζονται ειδικά μέτρα για την προστασία των παιδιών. Στις περισσότερες συζητήσεις μας ε, δεν το αναφέρουμε ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Αλλά χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση. Και όλα τα νομικά μας συστήματα, δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικέ διαδικασίες για τα παιδιά. Αυτό είναι σαφές. και πρέπει να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κάτι ακόμη. Πρέπει να μιλήσουμε για τα δεδομένα. Δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες. Και πρέπει να μας δώσουν πληροφορίες στα κράτη-μέλη. Το είπατε επανειλημμένως. Επομένως πρέπει να στραφούμε στα κράτη-μέλη και να το τονίσουμε αυτό. Λοιπόν, ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα και σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και σας ακούσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά σας και για τις εξηγήσεις σας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα τους επόμενους μήνες και φυσικά και στο νομικό μας πλαίσιο. Και Τώρα έχω να πω το εξή. Θα μου ζητηθεί να παρουσιάσω τα αποτελέσματα αυτού του εργαστηρίου στην Ολομέλεια, στην τελευταία συνεδρίαση. Θα το πράξω. Τώρα εσείς έχετε κάποιο διάλειμμα, κάποια λεπτά διάλειμμα, θα διακόψουμε μέχρι τις 4 παρατέταρτο και θα ξανασυναντηθούμε εδώ. Μπορείτε να μείνετε εδώ, μπορείτε να πάτε για καφέ και να ξανάρθετε. Στις 4 παρατέταρτο. Ευχαριστώ.